Dear colleagues, uh, we will start. Please sit down. Καλημέρα συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε αν έχετε την καλοσύνη. Good morning everybody. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω με την έγκριση της ε, ημερήσιας διάταξης. Αν συμφωνείτε όλοι με την ημερήσια διάταξη. Πολύ ωραία. Περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Τα έχετε τα πρακτικά στη διάθεσή σας. Αν υπάρχει κάποια ένσταση, όχι, τότε περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Είναι ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο να σας εκθέσω. Και γι' αυτό περνάμε ήδη στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι η φτώχεια και η προοπτική του φίλου. Μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Η συγκήτρια είναι η κυρία Αρένα, που θα κάνει την παρουσίασή της ακριβώς για το θέμα αυτής της έκθεσης. Και θα της δώσουμε αμέσως τον λόγο και μετά στους αρμόδιους των ομάδων. κυρία Ρένα παρακαλώ. Euh, Εντάχει, ήδη είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έγγραφο εργασίας. Συλλέξαμε επίσης κάποια σχόλια που διατυπώθηκαν. Σήμερα έχω την πρόταση έκθεσης που είναι διαθέσιμη για όλους τους κοιόδης εισηγητές που στρέφεται γύρω από δύο σημεία εντοπισμού του θέματος της φτώχειας, συσχετισμός μεταξύ φτώχειας και ισορροπίας επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, αλλά και η φτώχεια και ο συσχετισμό με την εργασία. Πολύ συχνά έχουμε την τάση να πιστεύουμε το θέμα τη φτώχεια είναι επιλημένο όταν έχει κανεί όλο στην εργασία. Δυστυχώ, όταν πρόκειται για τι γυναίκε, υπάρχει το θέμα τη διάκριση στην εργασία και υπάρχει βέβαια και το θέμα τη διάκριση στο μισθό. Λοιπόν, έχουμε πάντα την κατάσταση διάκρισης όσον αφορά την ισότητα των μισθών των συντάξεων που συνδέεται με το θέμα της καριέρας, που διακόπτεται η καριέρα των γυναικών, αλλά είναι και το θέμα ε, της ανασφαλούς, επισφαλούς εργασίας των γυναικών όταν ε, έχουν εργασία. Υπάρχουν κάποιες ε, συστάσεις οι οποίες διατυπώνονται, στρέφονται γύρω από κάποιους άξονες. Καταρχάς εντοπίζουμε και το εξή ότι τα φτωχά άτομα, κυρίως οι γυναίκες, παραδόξως πληρώνουν πιο ακριβά το κόστος κάποιων υπηρεσιών που τους παρέχονται σε σχέση με τα άτομα που έχουν περισσότερα χρήματα είναι παράδοξα, διότι όσο πιο φτωχοί είναι οι άνθρωποι πληρώνουν πιο ακριβά κάποιες υπηρεσίες. Το δεύτερο σημείο αφορά τη σχέση μεταξύ φτώχεια των γυναικών και τη φτώχεια των παιδιών θα πρέπει να βρούμε λύσεις, όταν βρίσκονται λύσεις για τις γυναίκες, βρίσκονται και λύσεις στο φαύλο κύκλο της φτώχειας και σε σχέση με τα παιδιά. Τρίτη έννοια είναι το θέμα ορισμός του νοικοκυριού και της ε, και καλυμμένης φτώχειας, κρυμμένης φτώχειας. Όταν ορίζουμε τα νοικοκυριά, καμιά φορά λησμονούμε να λάβουμε υπόψη την φτώχεια των γυναικών εντός του νοικοκυριού, εντός του σπιτιού μετά υπάρχει ε, η φτώχεια που συνδέεται από την οικονομική εξάρτηση, σχέση μεταξύ οικονομικής εξαρτήσεως και της βίας κατά των γυναικών και τέλος το θέμα της φτώχειας και του αποκλεισμού. Πολύ συχνά πρόκειται περί οικονομικής φτώχειας που διαφαίνεται, αλλά αυτή η οικονομική φτώχεια συνεπάγεται επίση και κοινωνική ούτως υπήν φτώχεια δυσκολίες, δηλαδή για πρόσβαση υπηρεσίες όπως είναι οι πολιτιστικές ε, υπηρεσίες ή άλλου είδους υπηρεσίες. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ένα τμήμα της εκθέσεως και περιμένω ανυπόμονα τυχόν τροπολογίες των συναδέλφων ούτω ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα το οποίο το θέλουμε να το προωθήσουμε όλους ιδιαίτερως το έχουμε στην καρδιά μας. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Ρένα. Και τώρα οι παρεμβάσεις των ομάδων. Ο κύριος Σεμπαστιαν παρακαλώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια. Κατά την άποψή μας έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι σημαντικότατο να σημειώσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της φτώχειας και του φίλου. Διότι οι γυναίκες πάντα έχουν περισσότερο, δέχονται συνέπειες περισσότερο της φτώχειας θα θέλαμε μήνυμα στον αυτό το σχέδιο κειμένου επί δύο θεμάτων που ήδη βρίσκονται στην έκθεση. Το πρώτο θέμα είναι η επιρροή των πολιτικών λιτότητας επί της αυξήσεως της στοχεία. κυρίως μεταξύ των γυναικών. Η συγγήτρια ήδη ανέφερε κάποια πράγματα για να αλλάξει η πολιτική της λιτότητας για μας είναι θέμα σημαντικότατο, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και σαφή καταδίκη των αλόγων πολιτικών που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη και διευθύνονται κατευθύνονται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο θέμα είναι το βασικό εισόδημα. Ε, είναι επίμαχο θέμα. Πιστεύουμε όμως ότι είναι η μόνη λύση για να αποφύγουμε τη φτώχεια, ε, να υπάρχει το ελάχιστο εισόδημα. Πιστεύουμε αυτή η έκθεση είναι ιδανικός χώρος να αναφέρεται αυτό. Τέλος, ε, θα θέλαμε να προσθέσουμε δύο θέματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Καταρχάς, η, ε, η δικαιοσύνη στον το κλίμα. Οι γυναίκες έχουν περισσότερο δέχονται τις συνέπειες του κλίματος. Θέλουμε δικαιοσύνη στον φάτο του κλίματος. Μετά, ανάπτυξη και αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί πάντα, σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΟΗΕ, στις αναπτυσσόμενες χώρες το επίπεδο της στόχιας ε, είναι μεγαλύτερο στις γυναίκες, αλλά οι γυναίκες είναι οι βασικοί παράγοντες της αλλαγής. Θα υποβάλουν σχετικέ τροπολογίες. Δεν θα υπάρχουν δυσκολίες να συμφωνήσουμε με την εισηγήτρια από αυτόν. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να την ευχαριστήσω, διότι θεωρούμε ότι έκανε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σουίκα, τέχετε τον λόγο παρακαλώ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Σε αυτή τη γνωμοδότηση διάβασα το σχέδιο εκθέσεως που συνέταξε η κυρία Αρένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Αρένα για τη δουλειά που κάνατε. Όπως γνωρίζετε, συζητούσαμε εκτενώς την ισότητα ανδρών και γυναικών. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα από όρο παρέχει από το 50-50. Όλοι το γνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι θέλουμε οι γυναίκες να αμείβονται εξίσου με τους άντρες για την ίδια εργασία, να εκπροσωπούνται εξίσου σε επιχειρήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια και στις θέσεις λήψης αποφάσεων. Και όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να εξαλειφθούν όσον αφορά τη συμφιλίωση επαγγελματική και ιδιωτική ζωής, αληθεύει ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερέ διακοπές στην καριέρα τους, στα διαδρομία του, είναι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μερική απασχόληση και αυτό επηρεάζει τη σταδιοδρομία τους και τις συνταξιοδοτικές τους εισφορές. Και αυτό επηρεάζει επίσης ε, και το πόσες γυναίκες ε, πέφτουν στην κατηγορία της φτώχειας. Δηλαδή η φτώχεια πλήττει περισσότερο τι γυναίκε. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, οι γυναίκε πρέπει να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην παιδεία. Ε, Μεγαλύτερε διευκολύνσει για τα παιδιά πρέπει να παρέχονται για να μπορούν να συνδυάζουν ιδιωτική και επαγγελματική ζωή. Όλοι πρέπει να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα στον αφορά το φύλλο και στην παιδεία, να μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα τμήματα τη αγορά εργασία οι γυναίκε και να μειώσουμε έτσι τη φτώχεια που τι πλήττει. Να τονίσω επίση τη διαβίω εκμάθηση και τη γυναική επιχειρηματικότητα πρέπει να υποστηρίζονται, διότι έτσι οι γυναίκε έχουν τι αναγκαίε δεξιότητε για να έχουν πρόσβαση σε θέσει εργασία υψηλή ποιότητα. Η ποικιλομορφία των σταδιοδρομιών θα πρέπει να προωθεί ώστε αντιμετωπίζονται οι κατατμήσει τη αγορά εργασία και όπω προαναφέρθηκε να προωθήσουμε την γυναική επιχειρηματικότητα όλο ιδιαίτερο. Ε, Όμω, το ΕΛΚ έχει κάποιες σοβαρές αμφιβολίες επί κάποιων παραγράφων όσον αφορά την αρχή της ε, επικουρικότητας, διότι κάποιοι τομείς δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές, όμως δεν μπορεί να θεσπίσει σχετική νομοθεσία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ελπίζω να το συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Κλείνοντας, να σας υπενθυμίσω ότι ήδη έχουμε τόνους ε, νομοθεσίας, καλύτερο θα ήταν να επιμείνουμε στην ορθή εφαρμογή αυτής. Το πρόβλημα είναι πάντα η εφαρμογή της νομοθεσίας. Και αν παραστεί αναγκαίων, χρειάζεται αναθεώρηση νομοθεσία στα κράτη-μέλη, αντί να θεσπίζεται νέα νομοθεσία. Βέβαια, αυτό είναι θέμα προσυζήτηση. Για μια ακόμη φορά, ευχαριστώ κυρία Αρένα για το έργο σας και ελπίζω στο τέλος να καταλήξουμε να έχουμε μια καλή έκθεση. Σας ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την εισηγήτρια για το έργο που επετέλεσε. Και ως γενικό θέμα, ζήτημα που θα ήθελα να τοποθετηθώ επ' αυτού, θέλω να πω ότι θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε σε όλες τις εκθέσεις που εγκρίνουμε το εξής αίτημα προς τα κράτη-μέλη ώστε να κάνουν μια πολιτική όσον αφορά τις επενδύσεις τους και τις δράσεις τους στην πολιτική ισότητα. Είναι μια απέτηση, μια διεκδίκηση που πρέπει να εντάξουμε σε όλες τις εκθέσεις. Να είναι σαφής ο στόχος, να γίνουν επενδύσεις σε ε, πολιτικές ισότητας και να μην γίνονται απλώς δαπάνες, θα γίνονται επενδύσεις και σε κάποια από τα εδάφια της έκθεσης είδαμε ότι γίνεται λόγος για την απέτηση να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί, τα κονδύλια. Πολύ καλό αυτό. Αλλά εγώ πιστεύω δεν είναι τόσο η ανάγκη αύξησης προϋπολογισμών και κονδυλίων, αλλά να δώσουμε προτεραιότητα στις πολιτικές ισότητας και στις πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αρνητική μεταχείριση βάρος των γυναικών και τη φτώχεια που υφίστανται οι γυναίκες. Γιατί διότι σε πολλούς από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών υπάρχουν προϋπολογισμοί και κονδύλια αλλά χωρίς προτεραιότητες για αυτό το θέμα. Ούτε είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν τις επιπτώσεις για τα κορίτσια και τις γυναίκες των δεινών που υφίστανται. Γι' αυτό λοιπόν αν πει κανείς να αυξηθούν, εγώ θα έλεγα όχι, να δοθούν προτεραιότητες και να έχουν στόχο την ισότητα Συμφωνούμε απόλυτα με την ανάγκη να υπάρχει νομοθεσία σε σχέση με τη γονεϊκή άδεια, μητρική άδεια και πατρική άδεια που έχει τροχοπεδηθεί, έχει παγώσει το θέμα από το Συμβούλιο και δεν φαίνεται ότι μπορούμε να πετύχουμε τίποτα στους επόμενους μήνες όσον αφορά τα ευέλικτα ωράρια που είναι ένα από τα θέματα και τα αιτήματα για να μπορέσουμε να ευνοήσουμε την απασχολησιμότητα των γυναικών Πιστεύω όταν κάνουμε λόγο για ελαστικά ωράρια πρέπει να γνωρίζουμε ότι για γυναίκες και άνδρες πρέπει να ισχύουν αυτά αν ισχύσουν διότι είναι ένα από τα θέματα που δυσχεραίνουν τη ζωή των γυναικών αυτά όταν έχουν παιδιά. Δεν είναι μόνο λοιπόν ένα πρόβλημα παιδιών, είναι, ε, των γυναικών, είναι πρόβλημα και γυναικών και ανδρών. Πρέπει να εργαστούμε λοιπόν υπέρ της ελαστικότητας για όλους. Και συμφωνούμε για την ανάγκη να υπάρχει ένα ελάχιστο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πράγματι ο κύριος Γιούνκερ πρόεδρος της Επιτροπής στο πρόγραμμά του για αυτή την κοινοβουλευτική θητεία συμπεριέλαβε την αναφορά σε αυτό το ελάχιστο εισόδημα ή ελάχιστο μισθό ευρωπαϊκό. Για τουλάχιστον εμείς ως ομάδα, η Άλντε και εγώ είχαμε ένα ε, συγκεκριμένο αίτημα αυτό για να προαχθεί το, η δέσμη μέτρων κοινωνικών μέτρων με αυτό. Και μια ερώτηση που υπευλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν θα αντιμετωπίσει στο μέλλον αυτή την έννοια του ελάχιστου μισθού εισοδήματος και υπάρχει ανάλυση, το αναλύεται αυτό το ζήτημα από πλευρά τους. Δίνουμε συνέχεια λοιπόν σε αυτό και θέλω να πω συμφωνούμε και με αυτό. Πιστεύω πρέπει να τονίσουμε περισσότερο την ανάγκη, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 10, στις, ε, στα προβλήματα των εφήβων. Νομίζω ότι σε σχέση με την ε, τις επενδύσεις ε, στην παιδεία και την εκπαίδευση οι, τα κορίτσια, οι έφηβες ε, που δεν έχουν καταρτιστεί και εκπαιδευτεί πάλι πρέπει να εντάσσονται στην ε, αρμοδιότητα υπό την αιγίδα της παιδείας και εκπαίδευσης και θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τους δείκτες αποτυχίας για τα παιδιά αυτά στις διάφορες περιφέρειες και επαρχίες σε κάθε χώρα, σε κάθε περιφέρεια με τα εκπαιδευτικά πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να γίνει μία ακόμα αναφορά στις πολιτικές εκπαίδευσης και παιδείας. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι είναι μια έκθεση αυτή που βαίνει πολύ καλά. Έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες. <clears throat> Θα ήθελα όμως να συγχαρώ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπιλμπάου. Η κυρία Βυσνιεύσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η φτώχεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυξάνεται συνεχώς και πραγματικά δεν γνωρίζει φύλλα. Βεβαίως είναι διαφορετικός ο τρόπος που πλήττει τα δύο φύλλα. Οι, οι στατιστικές δείχνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, πάνω από 25% των γυναικών αλλά και των ανδρών πλήττονται από τη φτώχεια παρόλο που πρόκειται για μια προηγμένη οικονομία. Το ίδιο ισχύει και για τον ε, κοινωνικό αποκλεισμό. Και υπάρχουν... Ε, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά τα οποία είναι μονογονεϊκά. Και στο σημείο αυτό δεν μπορούμε να παραμελήσουμε το γεγονός ότι στην κατηγορία αυτή κυριαρχούν οι γυναίκες οι οποίες ε, είναι, έχουν μονογονεϊκές οικογένειες πολύ περισσότερο από τους άνδρες. 60% είναι γυναίκες και μόνο 2% είναι άνδρες με παιδιά. Η φτώχεια είναι αιτία σημαντικών ε, παραμελήσεων στον κοινωνικό τομέα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσει τον αριθμό των ε, θυμάτων. Ε, η διέξοδος βεβαίω σε αυτό το φαύλο δεν μπορεί παρά να είναι μόνο η εκπαίδευση και η εργασία. Ε, πολύ συχνά οι γυναίκες ε, που βρίσκονται μονογονεϊκών οικογενειών πλήττονται επίσης και από την ε, ανεργία. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφώνεται ο χρόνος της εργασίας ελεύθερα. Ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών στην Ευρώπη θεωρεί ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμφιλειωθούν ο οικογενειακός βίος και η επαγγελματική ζωή. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επεξεργάζεται μια αναθεώρηση της οδηγίας που αφορά ακριβώς τη συμβατότητα αυτών των δύο τομέων. Και θα πρέπει να αποφεληθούμε αυτής της ευκαιρίας ούτως ώστε να εκπονήσουμε πιο ευέλικτα μοντέλα της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ούτε ώστε να υπάρχουν και τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις ε, συνθήκες ε, διαβίωσης και να πετύχουν κάποιους ε, επαγγελματικούς στόχους χωρίς να υπονομεύεται η οικογενειακή του ζωή. Ε, θα ήθελα να δώσω στην εισηγήτρια το εξή. Πώς ε, αντιλαμβάνεται την εξατομήκευση των ε, δικαιωμάτων στον κοινωνικό τομέα υπό την έννοια ότι το μοντέλο του νοικοκυριού δεν επιτρέπει κατ' ουσία να κρυθεί να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των γυναικών σε σχέση με την φορολογική επιβάρυνση. Ε, δεν θεωρεί ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε μοντέλο και να βάλουμε στην άκρη το μοντέλο του νοικοκυριού και να, ώστε να μπορούν να υπολογίζονται ατομικά τα εισοδήματα σε ατομική βάση. Και βεβαίω εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η κατάσταση των παιδιών ε, σε σχέση με την, α, σχέση με την οικονομική κατάσταση του πατέρα ή της μητέρας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την θαυμάσια αυτή έκθεση. Και θα ήθελα να θέσω τρία θέματα ιδιαίτερως. Το ένα αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, όπου ε, εδώ τονίζει το σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης όσον αφορά το θέμα της φτώχειας. Το ένα αφορά το, ε, το, σχολικό, το επίπεδο της, του σχολείου ε, και την ε, προσπάθεια να απαλληφθούν οι διακρίσεις κατά των γυναικών ούτως ώστε να συμμετέχουν περισσότερο και τα κορίτσια σε τομείς που τη δίνουν τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή. Ήδη από το σχολείο λοιπόν. Αλλά επίσης πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της διαβίου μάθησης και η δυνατότητα για τις γυναίκες να μπορούν να επανακαταρτίζονται και να αναλαμβάνουν ε, ευθύνες. Το δεύτερο αφορά το θέμα της επισφαλούς ε, εργασίας και της ε, ευελιξίας. Πρόκειται για δύο διακριτά θέματα τα οποία αναπτύσσεται εδώ και αφορούν την ισορροπία στην αφορούν την πρόσβαση στον στο χώρο εργασίας και την οικογενειακή ζωή, αλλά επίσης το θέμα της παροχής μεγαλύτερης προστασίας έναντι εκείνων που εργάζονται σε επισφαλείς ε, συνθήκες, γιατί είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των γυναικών που έχουν τέτοιου είδους επισφαλείς ε, συμβάσεις εργασίας. Και επίσης ε, για την παράγραφο 4 εδώ χρειάζεται να γίνει μια διευκρίνηση εν σχέση με τα δικαιώματα εξατομίκευσης στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ίσων δικαιωμάτων για τα δύο φύλλα. Αλλά, παρακαλώ, θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ γιατί πρόκειται για μια εξαίρετη έκθεση. Ωραία λοιπόν. Η κυρία Αρένα έχει το λόγο για να απαντήσει στις παρεμβάσεις που έγιναν σχέση με την έκθεσή της. Ωραία λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία επανέρχονται κυρίως στο θέμα της πρόσβασης στην εκπαίδευση και έλαβα γνώση το θέμα της, του θέματος της ε, διαβίου μάθησης που τέθηκε από τη συνάδελφα και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό δεδομένο το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε εδώ. Τώρα, το θέμα το οποίο τέθηκε από τη Ζορτή ιδιαίτερος στο θέμα της ε, ε, κλιματικής δικαιοσύνης και της αναπτυξιακής βοήθειας εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η έκθεση αυτή αφορά την φτώχεια των γυναικών στην Ευρώπη και δεν προσερκίζει το θέμα διεθνώς ε, της, πτώχειας, ε, της φτώχειας των γυναικών που θα απαιτούσε μια πιο περιεκτική και ευρία έκθεση. Βεβαίω αν διευρύνουμε το θέμα της φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο, ε, αυτό θα ενήχε το κίνδυνο ε, να μην ε, θα, έπρεπε να προσθέσει μάλλον να συμπεριλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι η έκθεση και να επεκταθεί πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ατομικών δικαιωμάτων, εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να πάμε περισσότερο προς την εξατομίκευση των δικαιωμάτων, αλλά δεδομένου ότι ε, υπάρχουν διάφορες απόψεις όσον αφορά την σύνθεση των δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, όσον αφορά την σταδιοδρομία υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την σταδιοδρομία τους γιατί για παράδειγμα αφησιάζουν το δικό τους δικαίωμα και το εκχωρούν στο σύζυγό τους ούτως ώστε αυτός να εκπληρώσει τη σταδιοδρομία τους. Ε, και το θέμα αυτό διαπλέκεται με το θέμα της στόχης, γιατί αν πούμε ότι μια γυναίκα δεν έχει πλέον δικαίωμα στη σύνταξη του συζύγου της, ε, τότε ε, θα βρεθεί πραγματικά σε μια κατάσταση φτώχεια στην ε, στιγμή της συνταξιοδότησης. Άρα θα πρέπει να γίνει μια βάθος ανάλυση του θέματος της εξατομίκευσης των δικαιωμάτων, να δούμε πού βρισκόμαστε. Αν έχουμε προχωρήσει αρκετά στο επίπεδο των χωρών μελών, ούτω ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε σε αυτή την λεγόμενη εξατομίκευση των δικαιωμάτων. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται σε κάθε χώρα για να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε στο κατά πόσο η εξατομίκευση τελικά οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτονόμηση ε, και οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών ή σε ορισμένες χώρες θα οδηγήσει ενδεχομένως σε μία ρήξη και θα κάνει πιο ευάλωτες τις γυναίκες ή πώς μπορεί να αντισταθμιστεί αυτός ο κίνδυνος. Για παράδειγμα, πολλές γυναίκες μιας γενιάς που σήμερα έχουν, ε, είναι γύρω στα 60 δεν έχουν πρόσβαση στο χώρο εργασίας γιατί αυτό το μοντέλο της κοινωνίας ήταν έτσι φτιαγμένο αλλά εάν ε, βεβαίως εξατομικευθούν τα δικαιώματα, τότε δεν θα έχουν πλέον κανένα δικαίωμα συνταξιοδότηση, γιατί δεν έχουν θεμελιώσει τέτοιο δικαίωμα ατομικά, σε ατομική βάση. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε οι χώρες μέλη θα πρέπει να αντισταθμίσουν αυτό το οποίο ε, θα τους έδινε το σύστημα συνταξιοδότησης στη βάση ενός ατομικού δικαιώματος το οποίο δεν έχουν κατοχυρώσει οι γυναίκες στην περίπτωση αυτή. Ε, και για, κατά τα άλλα περιμένω τις δικές σας τροπολογίες όσον αυτές τις διάφορες προτάσεις. Βεβαίως και το ζήτημα της ε, διασύνδεσης με ορισμένα δικαιώματα τα οποία ε, συνδέονται με το θέμα της ε, λιτότητας και πώς η λιτότητα ε, πλήττει ιδιαίτερο στην κατηγορία των γυναικών που είναι πιο εξαρτημένες από τις δημόσιες ε, υπηρεσίες. Αλλά περιμένω αυτές τις προτάσεις όταν συμπεριληφθούν ε, στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρένα. Θα ανοίξουμε ένα νέο γύρο παρεμβάσεων τώρα. Και είμαι σίγουρη ότι η κυρία Αρένα θα ε, είναι στη διάθεση των συναδέλφων για να ολοκληρώσει αυτό το διάλογο. Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά... Α, ναι, γιατί η προθεσμία υποβολή των τροπολογιών είναι 23 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα. Οριστοκο... Λίγη η προθεσμία αυτή. Στις 18 ε, θα ψηφιστούν ε, στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Μαρτίου, στην το επόμενο σημείο αφορά την εσωμάτωσή διάσταση του φίλου εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μίλναρ, η οποία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για την άριστη συνεργασία μεταξύ σχεδόν. Ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Οι συνάδελφοι ήθελαν να ασχοληθούν πολύ με το θέμα αυτό της λήψης υπόψη της διαστάσης του φύλου της εργασίας του Ευρωκοινοβουλίου. Συμφωνήσαν πενέα συμβαστικών τροπολογιών που συμπεριλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία της εκθέσεως. Δύο από αυτές, η 1 και η 3, έχουν σαν στόχο να υπογραμμίσουν τη σημασία του ρόλου των γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Συμβαστική τροπολογία 2 ζητά στο δίκτυο το αρμόδιο για τη λήψη υπόψη του φίλου να σκηνηθηθεί. Η 5, να, στον εσωτερικό κανονισμό να γίνουν αναγκαίε αλλαγέ για κάτι τέτοιο, ότι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ τη Επιτροπή Γυναικών και των Επιτροπών που δέχονται τις τροπολογίε συμβαστικέ 5 και 6 αντίστοιχα αφορούν τη σημασία που έχει πραγματικό εγχείρημα προσπάθεια να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου στι νομοθετικέ προτάσει. Συμβαστική 7. Η δεύτερη διάσταση τη διαστάσεως του φύλου λαμβάνοντας υπόψη την εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών στους τομείς πολιτικής και πόσο σημαντική είναι η κατάρτιση τη της του φύλου. Η οκτώ ζητά συγκεκριμένη δικασία για την έγκριση σχεδίων δράσεω για τη διάσταση του φύλου σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή και τελικά Συμβαστική Τροπολογία 9 υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η δημιουργία σωστού φορέα εποπτεία, ούτω ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι, οι προκαθοριστέντε. Το σύστημα ε, ε, για τη διάσταση του φίλου στο Κοινοβούλιο είναι κατακαιρματισμένο. Δεν υπάρχει διαδικασία αξιολόγηση, ούτε ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η έκθεση και οι συμπεφωνημένε συμβιβαστικέ συνετάχθησαν ούτω ώστε να υπάρχει πιο συνεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση και σχετικό σύστημα εργασία. Και είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που κάναμε τους τελευταίους μήνες και θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμμετείχαν συμπεριλαμβανομένες και της γραμματείας. Σας ζητώ λοιπόν να υποστηρίξετε συμβαστικές τροπολογίες ώστε να έχουμε ένα ισχυρό συνεκτικό συμπαγές κείμενο που θα υποβληθεί στην Ολομέλη. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. κύριε Μέλνα, γνωρίζετε ότι η ψήφιση αυτής της έκθεσης θα γίνει αύριο. Τώρα ξεκινάμε ένα γύρο παρεμβάσεων. Και θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚ η κυρία Πιετικάινεν, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ευχαριστώ την εισηγήτρια για την άριστη συνεργασία. Δεύτερον, όπως προαναφέρθηκε, είναι σημαντικό το, θέμα. Οι συμβιβαστικές και η έκθεση ακολουθούν άριστα την γραμμή του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, πρώτον, χρειάζεται η διάσταση του φίλου να λαμβάνεται υπόψη και από πλευράς ε, δημοσίων υπαλλήλων και από πλευράς εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Δεύτερον, χρειαζόμαστε και τα προγράμματα δράσεως, αλλά πρέπει να δοθεί σωστή συνέχεια και διευθυντικές δράσεις για να πετύχουμε το στόχο μας. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που συνεργαστήκαμε επί συγκεκριμένων δράσεων που πρέπει να αναλυθούν το Κοινοβούλιο. Να υπογραμμίσω δύο σημαντικότατα θέματα. Πρώτα απ' όλα, να λαμβάνετε υπόψη η διάσταση του φύλου στην αξιολόγηση συνεπειών, στις νομοθετικές διαδικασίες, αλλά και στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου και τις πολιτικές του. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σε θεσμικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλοι πόροι. Αυτό που υπογραμμίζουμε είναι ότι δεν βλέπουμε, αυτό που δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε και να δράσουμε. Άρα είναι κρισιμότατο να έχουμε τις αναγκαίες πληροφορίες και τους κατάλληλους πόρους για να το πετύχουμε αυτό. Από πλευρά ΣΕΛΚ. Συμφωνούμε με τη γενική γραμμή. Ίσως κάπου να έχουμε ξεχωριστές ψηφοφορίες. Το σημαντικό είναι ότι όταν γίνεται δια... μια, επιτρο... μια τέτοια συνεργασία μεταξύ επιτροπών πρέπει να συμφωνούμε των ενιών. Δεν είναι δύσκολο διότι έχουμε ήδη τις κατάλληλες πληροφορίες για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Έχουμε πολιτικές προτιμήσεις. Εγώ ίσως θέλω να αναφερθώ στην κυκλική οικονομία, την ευημερία των ζώων και να τα θέσω αυτά στο πλαίσιο της διάστασης του φύλου. Και νομίζω ότι θα είναι εποφελές για τις γυναίκες και για μας να έχουμε ξεκάθαρο πεδίο για αυτό που συζητούμε και να μην είναι πάρα πολύ ευρύ και να ξεχύνεται και σε άλλους τομείς πολιτικής που είναι εξίσου σημαντική για μας ως γυναίκες και ως άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά μια σημαντική έκθεση πιστεύω και ήταν πολύ θελκτικό με έλκυσε πολύ να εργαστώ για αυτή την έκθεση. Με μια συνεργασία μεταξύ όλων των εισηγητών σκιωδών και σε Ευχαριστώ για αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και τους βοηθούς μου και την, και την ε, Γραμματεία και την ε, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας βοήθησαν. Έχουμε ένα πολύ αξιόπιστο κείμενο, σχέδιο κειμένου για τη δράση που πρέπει να αναλυθεί για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ισότητας των φύλων από πλευράς Κοινοβουλίου. Εκεί έτσι εργαζόμαστε. Δεν λειτουργούν όμως πολύ καλά όπως θα έπρεπε τα πράγματα και αυτό θα κάνει τη διαφορά με την προσπάθεια που κάνουμε στην καθημερινή ζωή και δουλειά. Οι προτάσεις, ε, οι προτάσεις για την εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών, για την ε, πιστοποίηση των στελεχών, για την πιο αξιόπιστη δράση τους και την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση μετεξέλιξη των ατόμων που εργάζονται εδώ. Πώς μπορούν δηλαδή τα στελέχη αυτά να συλλέξουν πείρα και εμπειρίες και να πιστοποιηθούν αυτές σε σχέση με κατάρτιση ώστε στη σταδιοδρομία τους αυτά να ενδυναμωθούν. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμός μεταξύ φορέων για την ισότητα των φύλων, ιδιαίτερα συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών στην Επιτροπή Τρανς ξέρω ότι έχουν προχωρήσει, άλλες όμως όχι τόσο. Πρέπει οι βέλτιστες πρακτικές να εφαρμόζονται και να προαχθούν. Ένα άλλο θέμα, διαθεσμική συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου και η συμμετοχή των άλλων εταίρων στις βέλτιστες πρακτικές, οικουμενικά, είναι σημαντικό για μένα η προοπτική όχι μόνο για τις γυναίκες να τονιστεί, αλλά να τονίσουμε το ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για όλους, για όλους ανεξάρτητα από φύλο. Καμιά φορά επειδή είμαστε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών ξεχνάμε ότι είμαστε και μια Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, των φίλων, άσχετα αν είναι γυναίκες ε, ή άνδρες ε, εκείνοι στους οποίους απευθυνόμαστε. Και για τα σχόλια της κυρίας Αρένα για τα όσα είπε και για την έκθεσή μου για την ε, επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας και που πρέπει αυτό έτσι να εγκριθεί είναι μια έκθεση που έκανε λόγο για την γυναικεία μορφή, το γυναικείο πρόσωπο της φτώχειας. Όλα αυτά τα θέματα διασυνδέονται εγκάρσια, είναι αλληλένδετα. Το πώς θα εργαστούμε για την ισότητα των φίλων, την αξία που δίνουμε στο θεματολόγιο για την ισότητα, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Eh. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Πάνο έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και στην πρώτη συζήτηση που κάνουμε θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την εξαιρετική έκθεση από την κυρία Μίρναρ που θίγει ακριβοδίκαια τα προβλήματα και υποβάλλει και προτάσεις. Το είπαν και οι συνάδελφοι προλαλήσασες. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και για τις πολύ καλές συμβιβαστικές λύσεις τροπολογίες που προτάθηκαν. Έχουμε και μια σειρά τροπολογιών για τις συμβαστικές τροπολογίες, συνολικά για το ανοιχτό πνεύμα συνεργασίες που ήταν πολύ σημαντικό για μας, για τις ε, τροπολογίες για την ισότητα των φύλων, σημαντικό στοιχείο, δεσμευτικά να ληφθούν υπόψη από τι άλλε κοινοβουλευτικές επιτροπέ. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Θα καταθέσουμε μια προφορική τροποποίηση και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια ευρία αποδοχή για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Φορέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι είναι έξοχη έκθεση, σημαντικότατη για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Πιστεύω και για το θέμα της ισότητας των φίλων στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ εκ νέου την Αντζέλικα Βλίνερ Νίμπλερ και όλους τους συναδέλφους, του Σκιώδης που συνέβαλαν στην σύνταξη της εκθέσεως. Συντονίζομαι απολύτω με τη συνάδελφο του SND. Πιστεύω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά. Να υπογραμμίσω δύο σημεία που προστίθεται στα όσα αναφέρθηκαν. Εξίσου σημαντικά όμως. Στην έκθεση γίνεται λόγος για την ε, για το θέμα των ε, ΛΟΑΤ που μιλάμε ελάχιστα πρέπει να αναφέρουμε τέτοιου είδους ε, σχέσεις ως Ιταλίδα το λέω διότι συζητούμε καθυστερημένα μια βασική αναγνώριση της συμβίωσης πολιτικής, της συμβίωσης των ΛΟΑΔ και θα βοηθούσε να κινηθούμε, το συζητήσουμε και στο Κοινοβούλιο. Μετά και το θέμα της αξίας της δημοκρατίας ότιμης στο Κοινοβούλιο, της Συμπροεδρίας. Εδώ συζητούμε ποσοστώσεις. Χρειάζεται να υπάρχει η πολιτική εμπειρία της Συμπροεδρίας. Υποστηρίζουμε τις τροπολογίες συμβαστικές Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Εύχομαι αυτή η έκθεση να βοηθήσει να συντονίσουμε καλύτερα τις εργασίες όσον αφορά τη διάσταση του φύλου στο Κοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή και γενικά να λαμβάνει υπόψη η διάσταση του φύλου στις εργασίες μας. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Σας ευχαριστούμε. Κυρία Βυσνιέσκα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα από πλευράς μου να πω ότι πρώτα απ' όλα η τελευταία συζήτηση που διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά της βίας δηλαδή κατά εις βάρος των γυναικών κατά τη διάρκεια εκείνης της συζήτησης αποκόμισα την εντύπωση ότι η δική μου τοποθέτηση σε αυτή τη συζήτηση από τους συναδέφους λογοκρίθηκε. Δηλαδή λογοκρινόταν, λογοκρίνονταν τα όσα είχα πει από τους συναδέφους αυτής της Επιτροπής. Παρακαλώ να γίνονται σεβαστές οι απόψεις των άλλων. Άνθρωποι που έχουν άτομα που έχουν διαφορετικές απόψεις πρέπει να είναι σεβαστοί και οι απόψεις τους σεβαστές. Όσον αφορά αυτή την έκθεση, εδώ υπάρχει πάλι διαφορετική άποψη. Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν στην κοινοβουλευτική μας ε, ομάδα και να μην υποστεί επίθεση κανεί λόγω των διαφορετικών απόψεων που έχει. Πρέπει να δείξουμε κατανόηση. Η έκθεση, το σχέδιο έκθεση, επισημαίνει ότι η ένταξη της πολιτικής ισότητας των φύλων δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά το περιεχόμενο των τροπολογιών δεν είναι προς άλλη κατεύθυνση. Τι συμβαίνει ακριβώς εδώ λοιπόν η ιδέα της ισότητας των φύλων και των πολιτικών ισότητας των φύλων δεν σημαίνει για μένα ότι μπορούμε να έχουμε ποσοσ... στόχους που μπορούμε να ποσοστοποιήσουμε ή με ποσότητες να περιγράψουμε. Αυτό το οποίο για παράδειγμα εκπλήσει είναι η πρόταση ότι οι προτάσεις της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αυτόματα λέει και χωρίς να ψηφιστούν προς έγκριση θα εντάσσονται, λέει, στα κείμενα άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αναλύωτες οι προτάσεις αυτές. Πιστεύω ότι μόνο <clears throat> ότι όσοι πιστεύουν ότι μόνο μία κοσμοθεωρία είναι σωστή είναι χαρακτηριστική κατάσταση για τους κομμουνιστές το πρώην καθεστώς του κομμουνισμού ως κρατικό καθεστώς. Η ανάλυση των στοιχείων από το 2014 είναι ιδιαίτερα επιλεκτική και καταδεικνύει σαφώς το έγγραφο ότι οι τροπολογίες που αφορούν το θέμα της ένταξης της πολιτικής ισότητας των φύλων καταδεικνύεται αυτό σε 85% όσον αφορά την υποστήριξη ακριβώς των γυναικών αυτές οι τροπολογίες τι κάνουν. Έχουν την προσθήκη γυναίκα ή μ, όταν πρόκειται για γυναίκες. Με αυτή την προσθήκη λειτουργούν. Και θέλω να επισημανώ ότι η οταν προκειται για γυναικες καταδεικνύει και κάτι άλλο. Ότι δεν υπάρχει διασύνδεση ή αλληλεξάρτηση μεταξύ παρουσίας γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και της αποτελεσματικότητας της δουλειάς ε, ως ατόμων ε, των όσων συμμετέχουν σε αυτά τα συμβούλια. Με άλλα λόγια, κατά τη στιγμή της ανάλυσης η Επιτροπή ΕΝΒΗ, η, Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε γυναικεία ε, ήταν στην πλειοψηφία ε, από γυναίκες συναπαρτιζόταν. Πάμπολες εκθέσεις ε, υιοθετήθηκαν αλλά μόνο τρεις είχαν σχέση με την πραγματική κατάσταση των γυναικών. Και όλα αυτά τι δείχνουν Μία εισηγήτρια μόνο ήταν γυναίκα και μάλιστα προερχόταν από τη δική μας ε, κοινοβουλευτική επιτροπή. Δηλαδή αυτό το σχέδιο έκθεσης είναι υπέρ της ένταξης της πολιτικής ισότητας των φίλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά για να κοιτάξουμε γύρω μας, 8 άνδρες και 66 γυναίκες ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής μας. Ε, δεν είναι υπέρ της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το ίμιση δηλαδή από άνδρες και κατά το ίμιση από γυναίκες. Θα πρέπει κανείς να εμπλέκεται σε, ένα έργο όταν ενδιαφέρεται να εμπλακεί σε αυτό και να συνεισφέρει σε αυτό και όχι με ποσόστοση 50-50% να ισοπεδώνουμε τα πράγματα και έτσι να επιβάλλουμε μια στρατηγική. Πρέπει να επανεξετάσουμε λοιπόν τη στρατηγική μας και να καταλήξουμε σε μια νέα ε, αναθεωρημένη στρατηγική επί του θέματος γιατί διαφορετικά η μόνη ομάδα η ομάδα των γυναικών που η κατάστασή της ε, θα βελτιωθεί ε, μόνο οι εισηγήτριες στην Επιτροπή μας θα ασχολούνται και θα είναι αυτή η ομάδα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και σε αυτό το Κοινοβούλιο είναι αυτονόητο ότι σεβόμαστε τις ιδέες των άλλων και που είναι διαφορετικές ιδέες από ιδέες άλλων συναδέλφων. Και κάτι άλλο επίσης. Η δημοκρατία σέβεται την πολιτική διαφωνία και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συζητούμε, κάθε να εκθέτει τις απόψεις του ελεύθερα και να λέμε ότι η δημοκρατία είναι πλειοψηφικά η θέση των όσων εκφράζονται, όπως στη δική μας Επιτροπή. Τον λόγο έχει η κυρία Μόντι ε, Ευχαριστώ πολύ σε αντίθεση με αυτά που υπόθηκαν, ίσως θα κινηθώ. Απευθύνομαι όλος ιδιαιτέρως στη συνάδελφο αναφέρθηκε υπολογής 5 και 6. Ευπρόσδεκτο το ότι οι τροπολογίες για τον προπολογισμό ελαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου αναφέρεται και είναι σημαντικό. Αφορά τα πρακτικά μέτρα προσλήψη να γίνει ένας προϋπολογισμός και αποτίμηση μετά τις δράσεις. Να λάβουμε υπόψη μάλλον το, το πώς βάλει υπόψη η διάσταση του φύλου. Και με σωστή προσέγγιση θα πετύχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα... Ποιος? Head, Jag hade inte tänkt uttala mig, men jag känner ändå... Jag har varit här i tolv år nu i Europaparlamentet och eh, har ju sett... Είναι 12, εδώ και 12 χρόνια με μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρακολούθησα την εξέλιξη, τη μη εξέλιξη των ε, θεμάτων που σχετίζονται με την ισότητα των γυναικών. Δηλαδή σημειώνονται πρόοδοι αλλά πολύ, με πολύ αργό ρυθμό. Υπάρχουν πολύ λίγες ε, γυναίκες που κατέχουν υψηλά αξιώματα. Και το θέμα αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι στη βάση όλων των ε, θεμάτων προσεγγίσουμε τόσο στο πλαίσιο της Επιτροπής αλλά και των άλλων Επιτροπών. Δείτε τη συνθήκη της Λισαβόνας, δείτε τις ευ... όλες τις ευθύνες που έχουμε στη βάση της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί μια πλήρης ισότητα ευκαιριών, όμως αυτό δεν υπάρχει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπερασπιστούμε την ισότητα των φίλων σε όλες τις επιτροπές και επίσης κόλπους των πολιτικών ομάδων. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα δέκτυο υπευθύνων ατόμων σε όλες τις επιτροπές. Αλλά κυρίως θα πρέπει περισσότεροι άνδρες να συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις. Εμένα με θλίβει το γεγονός ότι κάθε φορά που γίνεται μια συζήτηση για την ισότητα των φίλων δεν υπάρχουν παρά μόνο γυναίκες που ενδιαφέρονται πόσοι άντρε παρίστανται ε, αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, για παράδειγμα. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να λύσουμε το πρόβλημα της ισότητας αν δεν υπάρξουν περισσότεροι άνδρες που να συμμετάσχουν σε αυτή την εργασία και που να κατανοούν ότι είναι ένα θέμα σημαντικό για ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο με ανησυχεί. Ε, υπάρχει, αυτό το πράγμα με ανησυχεί να βλέπω τη βραδύτητα με την οποία εξελίσσονται οι εργασίες εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Αγγέλικα Μέλιναρ έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα τα καλά σας λόγια και την υποστήριξή σας και ελπίζω ειλικρινά ότι θα αντικατοπτριστούν όλες αυτές οι θέσεις στην αυριανή ψηφοφορία και στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άρα ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της σημερινής συζήτησης. Θα περάσουμε στο σημείο 8 και θα δώσω αμέσως ε, το λόγο στην Μιχαέλα Ζοντροβά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω την γνωμοδότησή μου όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας ε, για την διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Ήθελα να τονίσω ότι οι γυναίκε στην Ευρώπη ακόμα ε, αντιμετωπίζουν διακρίσει στην αγορά εργασία. Οι γυναίκε είναι κυρίω εκείνε που έχουν την πρώτη ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών και των οικοκυριό και την οικογένεια. Και αυτές οι ευθύνες έχουν άμεση επέπτωση και άμεσο αντίκτυπο στις σταδιοδομίες των γυναικών και επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση και, τις συνθήκες, ε, και τα οικονομικά των γυναικών. Είναι ότι σε όλες τις χώρες μέλη έχουν εφαρμοστεί, έχουν μεταφερθεί οδηγία, έχει μεταφερθεί οδηγία στην εθνική νομοθεσία. Αλλά η νομοθεσία από μόνη της ε, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ισότητα. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα όσον αφορά τους κατάλληλους ορισμούς για το θέμα των διακρίσεων υπάρχουν πολλά ελλείμματα όσον αφορά τη συγκέντρωση δεδομένων και υπάρχει και σε ευαισθητοποίηση των γυναικών, η συνειδητοποίηση της κατάστασής τους. Ε, ε θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και ένας ε, μηχανισμός αντιμετώπισης περιπτώσεων διάκρεσης Και ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαφορές ε, στις ε, αποδοχές μεταξύ των δύο φύλων. με ενδιαφέρον τη συνεργασία με το Σιώδη και θα είμαι ευτυχής να υποστηρίξω τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα αμέσως το λόγο στην κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν μπορώ παρά να πω καλά λόγια στην εισηγήτρια σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική σας ε, δουλειά μέχρι στιγμής και θα ήθελα ιδιαίτερα να σε επισημάνω κάτι το οποίο θεωρώ πολύ θετικό, την επισήμανση των προβλημάτων που έχουν οι χώρες όσον αφορά ε, στην ερμηνεία του όρου των πολλαπλών ε, διακρίσεων. Δεν πρέπει να δούμε την οδηγία απομονωμένα αλλά σχέση με την οδηγία για την ισότητα ευκαιριών του 2006 και θα πρέπει να δούμε τις δύο οδηγίες συνολικά και θα πρέπει να ε, εξετάσουμε τα, τις αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή της έκθεσης σαν Ζαμπόρσκα γιατί βλέπουμε ότι πάντοτε προβάλλονται ενδιαφέρουσες ιδέες αλλά τελικά χωλένουν πάρα πολύ τα πράγματα στο πεδίο της εφαρμογής. Ε, για παράδειγμα, η προηγούμενη έκθεση κατάρτιση προπολογισμού ε, για την πολιτική των ε, φύλων. Εάν δούμε τα παραδείγματα όπου όταν εφαρμόζεται έχουμε τόσο θετικά αποτελέσματα, για παράδειγμα στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης, μέτρα τα οποία αφορούν την ε, μερική εργασία και ήταν μέτρα τα οποία πραγματικά ήταν εξαιρετικά σημαντικά γιατί οι επιπτώσεις της κρίσης ε, για τις γυναίκες ήταν λιγότερο ορατές από ό,τι για τους άνδρες. Και αν δούμε τα θέματα αυτά υπό το πρίσμα αυτής της ε, θεματολογίας θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο των ε, διακρίσεων που υποκρύπτονται εδώ. Δεν... Ε, και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν θα πρέπει πάντοτε να εξετάσουμε πολιτικά μέτρα όπως αναφέρεται και στις εκθεσίες και από την έννοια αυτή χαίρομαι πάρα πολύ για την μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλε παρεμβάσει. Έχουμε τη δυνατότητα επίση να έχουμε την παρουσία της Επιτροπής. Αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα γίνεται, η συζήτηση, γίνεται μια συζήτηση στην Επιτροπή απασχόληση και άρα λοιπόν η Επιτροπή δεν παρίσταται εδώ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες 23 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα. Ωραία λοιπόν και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο που αφορά την παρουσίαση της ε, μελέτης για την ανάλυση των πολιτικών κομμάτων και για την, όσον αφορά την ισόρροπη εκπρόσωπη των φύλων μετά τις εκλογές του 2014. pense que πώς είμαστε έτοιμοι και έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να σας μιλήσω για τη μελέτη μας, λέει κύριε Μακάκαρ, που ανετέθη από αυτή την Επιτροπή. At, um... Μας ζητήθηκε να εξετάσουμε γιατί υπάρχουν λιγότερες γυναίκες ευρωβουλευτές από άντρες εν συγκρίση με τις πρώτερες ευρωεκλογές μάλιστα. Η μελέτη μας ανέλησε τα πολιτικά κόμματα και ανεξαρτήτους υποψηφίους και πολιτικές για την ισορροπία των φύλων στο Ευρωκοινοβούλιο που προήλθε από τις τελευταίες ευρωεκλογές. Είμαι Κέιτι Μακράκεν, ε, διευθύνω το Opsit Research που εδρεύει στο Λονδίνο. Μας ζητήθηκε να κάνουμε τα εξής. Εξού και οι στόχοι της μελέτης που επεκτάθησαν κάπω. Προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε εν γέννη γιατί υπάρχουν λιγότερες γυναίκες ευρωβουλευτέ από ότι άντρε. Θέλαμε να κατανοήσουμε ποια είναι η συνέπεια των διαφορετικών εκλογικών συστημάτων των κρατών μελών. Πώς επηρέασε τις πιθανότητες των γυναικών να εκλεγούν. Διερευνήσαμε και πώ οι ποσοστώσει λειτουργούν ή δεν λειτουργούν. κυρίω πώς οι ποσοστώσεις επηρεάζουν γενικά το θεσμικό εκλογικό πλαίσιο. Μπορεί σε ένα πλαίσιο να λειτουργούν καλά οι ποσοστώσεις και όχι σε άλλο. Σε ποιο πλαίσιο δίνουν αποτελέσματα οι ποσοστώσεις, σε ποιο όχι. Θέλαμε να δούμε τις συνέπειες που έχουν οι ποσοστώσεις όσον αφορά τη συμπεριφορά των κομμάτων. Αξιωματούχους των κομμάτων, πολιτικές των κομμάτων κλπ. Πώς επηρεάζονται. πώ επηρεάζονται οι πεπιθήσεις των υποψηφίων και η συμπεριφορά του. Θέλαμε να καταλάβουμε επίσης εν γέννη ζήτηση και προσφορά και πώς επηρεάζει αυτό την εκλογή των γυναικών ως ευρωβουλευτές. Ποια ζήτηση υπάρχει γυναίκες ευρωβουλευτές. Θα διατρέξω τις χρησιμοποιηθήσεις μεθόδους. Εξετάσαμε τα διάφορα εφιστάμενα κείμενα και στοιχεία για την προσφορά και ζήτηση για γυναίκες υποψηφίους και την τελική τους εκλογή. Διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα σε νέα κράτη-μέλη, ήρθαμε σε επαφή με ευρωβουλευτές και κροσόπους πολιτικών κομμάτων, με οργανώσεις γυναικών. Συναντηθήκαμε με υπευθύνου για την επιλογή υποψηφίων στα διάφορα κράτη-μέλη. Ήρθαμε σε επαφή και με ευρωβουλευτές και γυναίκες ευρωβουλευτές και υποψήφιες. Πολύ πρωτότυπη έρευνα. Προβήκαμε σε μια ποσοτική ανάλυση. Εξετάσαμε μια ευρεία βάση δεδομένων που αφορούσε γυναίκες υποψήφιες τελευταίες εκλογές. Στην ανάλυση εξετάσαμε τα διάφορα χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Χώρα καταγωγής, χώρα έδρας μάλλον, κόμμα, ήταν ανοιχτό στο σύστημα ή με λίστα εξελέγησαν, ήταν υποψήφιες. Πόσο ήταν καινούριε υποψήφιες ή όχι, παράγων φύλου κλπ. Κάναμε διάφορες αναλύσεις. Είχαμε στατιστικά στοιχεία περιγραφικά, κάναμε επισκόπηση του αριθμού των υποψηφίων που πέτυχαν, των γυναικών που πέτυχαν, εξελέγησαν, το είδος του εκλογικού συστήματος, κάναμε και αναδρομική ανάλυση. Υπολογίσαμε την πιθανότητα μία υποψήφια να εκλεγεί κατά πόσο οι άνδρες υποψήφοι ήταν πιο πιθανό να εκλεγούν από τις γυναίκες, ανάλογα με το σύστημα και τις ποσοστώσεις που χρησιμοποιούσαν. Ταχεία επισκόπηση είναι αυτή, θα γνωρίζετε όλοι το γράφημα, τα αποτελέσματα των εκλογών του 2014. Μόνο 2% αύξηση είχαμε στον αριθμό των γυναικών ευρωβουλευτών. Απογοήτευσε πολλούς αυτό. Είδαμε ότι τα αριστερίζοντα κόμματα είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών ευρωβουλευτών. Η Συμμοσπιακή Ομάδα της ε, Νοτικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς είχε το υψηλότερο επίπεδο. Ακολούθησε μετά η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, οι Ευρωπαϊκοί Συντηρητικοί και οι Μεταρρυθμιστές είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών ευρωβουλευτών. Βλέπετε στο γράφημα αυτό τις διαφορές σε ποσοστά γυναικών ευρωβουλευτών κατά κράτος μέλος και σύγκριση μεταξύ 2009-2014. Εδώ βλέπετε τα ποσοστά των πολιτικών ομάδων. Βλέπουμε τις γυναίκες ευρωβουλευτές στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Τι διαπιστώσαμε από τις μελέτες τις άλλες και τα κείμενα. Υπάρχει, υπάρχει τεκμηρίωση σχετικά με το γιατί είναι λιγότερες γυναίκες ε, πολιτικοί στην αντιπροσωπευτική ε, πολιτική αν θέλετε από τους άντρες. Παρουσιάζουμε κάποια από τα πορίσματα. Δεν υπάρχουν δεσμευτικέ διατάξει ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενθάρρυνση των πολιτικών κομμάτων ή των κατών μελών να θεσπίσουν ποσοστώσει ή άλλα θετικά μέτρα για να επιτυγχάνει την εξορρόπηση των φύλων. Οι ερευνητέ αναφέρονται εκτενώ την προσφορά και τη ζήτηση και τους σχετικούς παράγοντες. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από τον αριθμό των γυναικών ευρωβουλευτών, παράγοντες προσφοράς, πόσες γυναίκες δηλαδή υποψήφοι είναι διαθέσιμες ε, για εκλογή. Συμπεριλαμβάνονται εδώ στοιχεία όπως έλλειψη μοντέλων ε, στην πολιτική γυναικών που αποτελούν πρότυπο. Η νοτροπία ευνοεί ε, τους άντρες αρνητική προβολή στα ΜΜΕ. Κάτι που αποθαρρύνει τις γυναίκες να θέλουν εμπλακούν στην πολιτική. Αυτό επηρεάζει την ε, προσφορά γυναικών που θέλουν υποψήφιες. Ζήτηση για γυναίκε υποψήφιου. υποψήφιες μας, συγγνώμη, στα συστήματα με κλειστή λίστα, τα κόμματα θα πρέπει να θέλουν συμπεριλαμβάνουν τις γυναίκες στη λίστα. Διότι σε αυτά τα συστήματα, τα κόμματα ελέγχουν πόσε γυναίκε θα μπουν στη λίστα. Και θα πρέπει να θέλουν να βάλουν στις λίστες ε, προτεραιότητε γυναίκε γυναίκες για πολύ υψηλά αξιώματα. Στα ανοιχτά συστήματα πρέπει να βοηθηθούν οι γυναίκε στους ψηφοφόρου για να κερδίσουν έδρε. Και περισσότερο σε αυτό το σύστημα, όπω και στα άλλα, αλλά περισσότερο εδώ, είναι πιο δύσκολο να πετύχουν τη θέση οι γυναίκε. Και ίσω και η κοινωνία στηρίζει λιγότερο τι γυναίκε στην πολιτική. Υπάρχει επικρατή παράδοση με βάση το φύλλο. Η τεκμηρίωση αυτό έδειχνε. Θέλαμε να δοκιμάσουμε αυτές τις θέσεις και τις θεωρίες. Αν Δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες του πίνακα. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα στοιχείων. Περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών βλέπετε. Στο άκρο δεξιά στη στήλη βλέπουμε πιθανότητες ανδρών και γυναικών υποψηφίων για τις εκλογές του 2014. Οι υποψήφοι τι πιθανότητα είχαν. Ποιες οι πιθανότητες των γυναικών να συγκρίσει με τους άντρες. Είναι πάνω από έναν υπέρ των γυναικών, κάτω από έναν υπέρ των ανδρών οι πιθανότητες. Βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορα συστήματα. Είδαμε αν είναι σύστημα με λίστα, ανοιχτό σύστημα, ανάμειξη των δύο, τι είδους ποσοστώσεις χρησιμοποιήθηκαν, αν δεν υπήρχαν καθόλου και όταν υπήρχε ποσόστοση. Βλέπαμε αν ισχύει για όλη τη λίστα, μέρος της, λύση, της λίστας κλπ. Πώς εφαρμοζόταν η ποσόστοση με άλλα λόγια. Εξετάσαμε διάφορες μεταβλητές. Οι λεπτομέρειες στην έκθεση. Συνοψίζω τον πίνακα. Γενικά. Υπάρχει θετική επιρροή όσον αφορά τι πιθανότητε εκλογή γυναικών όταν χρησιμοποιούνται ποσοστώσει. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Υπάρχουν πολλέ διαφορέ μεταξύ κρατών μελών και πώ επηρεάζουν ποσοστώσει στην κατάσταση στα κράτη-μέλη. Όταν χρησιμοποιήθηκαν ποσοστώσει, είδαμε ότι εν γέννη αυτό ήταν ευνοϊκό για τι γυναίκε. Είχαν περισσότερε πιθανότητε να εκλεγούν. Άρα, συνεπώ, δεν είδαμε αρνητική συνέπεια χρήση ποσοστώσεων δεν μειωνόταν οι πιθανότητε των γυναικών να εκλεγούν από τη στιγμή που έθεταν την υποψηφιότητά του, υπέβαλαν υποψηφιότητα. Για χώρε που χρησιμοποιούσαν κλειστέ λίστε, τα σχετικά συστήματα, κλειστά συστήματα εκτό από Γαλλία και Ισπανία, οι γυναίκε ήταν πιο πιθανό να εκλεγούν. Αυτό ίσχυε όλο ιδιαίτερω για Ρουμανία και Σλοβακία. Παρά το ότι είχαν χαμηλότερα ποσοστά υποψηφίων, γυναικών υποψηφίων εν πρώτη, καταρχά. Τι δείχνει αυτό ότι σε κλειστά συστήματα τα κόμματα ίσως να προθούν τις γυναίκες ούτως ώστε να αντισταθμίσουν το χαμηλό αριθμό γυναικών που είναι υποψήφιες. Παρά τα αυτά, οι γυναίκες είναι πολύ λιγότερες ως ευρωβουλευτές που προέρχονται από αυτές τις χώρες. Άρα, ποιο είναι το επιχείρημα. Λιγότερες γυναίκες υποψήφιες είναι ο λόγος για τον οποίο εκλέγονται και λιγότερες γυναίκες τελικά. Η χρήση των ποσοστώσεων φαίνεται να συνδέεται με ίση πιθανότητα εκλογής ανδρών και γυναικών στα συστήματα με κλειστή λίστα, όταν δεν χρησιμοποιείται ποσόστοση, οι γυναίκες τελικά είναι πιθανότερο να εκλεγούν. Um, now this is, this is important because many, uh, Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πολλοί επιχειρηματολογούν λέγοντας λέγοντας ότι υπάρχει αντίληψη ότι ίσως οι γυναίκες δεν θα είναι δημοφιλείς με τους ψηφοφόρους. Και σχετικά με αυτό το επιχειρήμα αναφέρεται ότι οι γυναίκες ίσως δεν έχουν επαρκή εμπειρία ούτως ώστε να θεωρούνται επάξιες υποψήφιες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό δεν αληθεύει. Από τη στιγμή που υποβάλλουν υποψηφιότητα έχουν, έχουν ίσες πιθανότητες οι γυναίκες είναι πιο, ίσως και πιο δημοφιλής, είναι εξίσου δημοφιλής, ίσως πιο δημοφιλής από ότι τους άντρες όσον αφορά το εκλογικό σώμα. Σε μικρά συστήματα η χρήση των ποσοστώσεων είναι υποφελής για τις πιθανότητες των γυναικών να εκλεγούν. Όταν δεν υπάρχει ποσοστώσεις, οι γυναίκες έχουν πιο λίγες, πολύ πιο λίγες πιθανότητες να εκλεγούν εν συγκρίση με τους άντρες. Όταν συγκρίνουμε άντρες και γυναίκες υποψηφίους, σαν άτομα, και πόσες πιθανότητες έχει το κάθε άτομο να εκλεγεί. Υπάρχει θετική συνέπεια τη χρήση των ποσοστών στην γυναίκε στα ανοιχτά συστήματα, βελτιώνεται η πιθανότητα να εκλεγούν. Ήδη αν έχουν περισσότερε πιθανότητε να εκλεγούν σε αυτά τα συστήματα από ότι άντρε, με την ποσόστοση αυξάνονται αυτέ οι πιθανότητε. Οι γυναίκε βέβαια είναι δημοφιλεί ω υποψήφιε. Κάναμε και κάποια ανάλυση αναδρομική, κάναμε προβολέ προ το παρελθόν, να δούμε πώ Άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τις πιθανότητες εκλογής των γυναικών. Είδαμε διάφορα. Μεταβλητές που προανέφερα. Αλλά και κατά πόσο είναι παλιές υποψήφιες, γνωστές. Πώς επηρεάζεται, ποια είναι η θέση του στη λίστα. Τι είδαμε λοιπόν την ανάλυση θετική τάση προς τις γυναίκες στα ανοιχτά συστήματα. Αυτό μας εκπλήσει όλος ιδιαίτερος. Επίσης εξίσου και πόσο είναι γνωστές αυτές οι γυναίκες, ήταν και παλιά υποψήφιες. Όταν είναι γνωστές και έχουν επανεκλεγεί είναι πολύ πιο πιθανό να εκλεγούν ξανά. η ποσόστοση επηρεάζει την πιθανότητα να εκλεγούν οι γυναίκες στα ανοιχτά και στα κλειστά συστήματα. Και αυτό σε συνάρτηση εμά με τα βλήτες. Στα συστήματα με ανοιχτές λίστες οι προβολές έδειξαν ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εκλεγούν από τους άντρες ανεξάρτητα αν υπάρχει ποσόστοση υπέρ των γυναικών ή όχι. Το επαναλαμβάνω. Ποιο είναι το βασικό μάθημα. Οι γυναίκες είναι δημοφιλεί όσον αφορά το εκλογικό σύστημα, όταν οι εκλογείς μπορούν να προτιμήσουν ατομικά συγκεκριμένο υποψήφιο, τότε μπορούν να, πιθανότερο είναι να εκλέξουν γυναίκα. Προτιμούν τι γυναίκες σε ατομικό επίπεδο. Σε πολλά κράτη-μέλη, οι γυναίκες ω υποψήφιες έχουν περισσότερη πιθανότητα να εκλεγούν εν συγκρίση με τους άντρε. Τα πολιτικά κόμματα με τα κλειστά συστήματα ίσως να προωθούν τις γυναίκες υποψηφίους και έτσι αυξάνεται η πιθανότητα εκλογής τους εν συγκρίση με, άλλες, με άλλους υποψηφίους στα κλειστά συστήματα. Ποιο είναι το συμπέρασμα από την έρευνα. Ότι ο, ο μικρός αριθμός των γυναικών ευρωβουλευτών οφείλεται ότι είναι λιγότερες γυναίκες υποψήφιες. Αλλά όταν είναι υποψήφιες έχουν καλές πιθανότητες να εκλεγούν. Πρέπει να βάζουν περισσότερες γυναίκες υποψηφιότητα. Αυτό είναι το συμπέρασμα. findings from our case studies and we did... Λοιπόν, ερευνήσαμε την κατάσταση σε 9 κράτη-μέλη. Μιλήσαμε με ευρωβουλευτέ, εκπροσώπου των κομμάτων και ομάδε γυναικών, όπω ανέφερε επανειλημμένα. Στα πολιτικά κόμματα υπάρχει πεποίθηση ότι στάση έναντι των θετικών δράσεων όπως είναι οι ποσοστώσεις, η τοποθέτηση είναι θετική. είναι αντιλήψεις παγιωμένου εντός του κόμματος που διαμορφώνονται και παραμένουν. Και ποιες είναι αυτές. Λένε κάποιοι ότι είναι κατά ποσοστώσεων. Γιατί το λένε αυτό. Λένε ότι ε, οι εκλογές πρέπει να βασίζονται στα προσόντα και σε τίποτα άλλο. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα για αυτούς που είναι αντίθετοι. Οι αριστεροί και οι πράσινοι θέλουν θετικά μέτρα όπως είναι οι ποσοστώσεις. Και οι συντηρητικοί και οι δεξιοί δεν θέλουν τέτοια μέτρα. Τούτο λεχθέντος όμως μεταξύ συντηρητικών και δεξιών κομμάτων υπήρχε η πρόθεση να βελτιωθεί η ισορροπία των φίλων και να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες, περισσότερες γυναίκες να είναι υποψήφιες. Δεν θέλαν όμως να θεσπίσουν θετικά μέτρα όπως προσωστώσεις. Υπάρχει ποικιλία προσεγγίσεων όσον αφορά την κατάρτιση των καταλόγων των κομμάτων, την κατάρτιση της λίστας. Κάποια κόμματα χρησιμοποιούν ποσοστώσεις, κάποια άλλα όχι. Κάποιε χώρε θεωρούν ότι οι ποσοστώσει δεν χρησιμοποιούνται διότι οι γυναίκε έχουν ίσε ευκαιρίε με του άντρε να εκλεγούν. Άρα δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Σε κάποιε περιπτώσει, όταν υπάρχει νομική πρόβλεψη υποχρεωτική για ποσοστώσει και επιβάλλεται στα κόμματα για την κατάρτιση του καταλόγου τη λίστα. τότε καμιά φορά τα κόμματα προσπαθούν να πετύχουν το ελάχιστο απαιτούμενο και δεν ξεπερνούν το όριο. Και αν είναι χαμηλή ποσόστοση, αυτή η χαμηλή ποσόστοση δεν βοηθά την εξισορρόπηση των φύλων. Η αποτελεσματικότητα στρατηγικών για τη βελτίωση τη ισορροπία των φύλων μειώνεται πολύ από τα εκλογικά συστήματα που ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα. Δυσχερέστατο για μα λοιπόν να συναγάγουμε συμπεράσματα. Να βρούμε ποια είναι η λύση που πρέπει να εφαρμοστεί καθολικά για να βελτιωθεί η ισορροπία των φύλων όσον αφορά του ευρωβουλευτέ που προτείνονται. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι έχουν θετικά αποτελέσματα οι ποσοστώσεις. Είναι σαφές αυτό τα στοιχεία. Πολλοί εκπρόσωποι οργανώσεων γυναικών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και κάποιοι εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, δηλαδή οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση της λίστας του κόμματος, διατείνονται ότι συστήματα με κλειστό ε, ε συστήμα, με κλειστό κατάλογο Party list Εάν το εκλογικό σύστημα είναι ανοιχτό, οι γυναίκες ίσω εργάζονται πιο σκληρά από τους άντρε για να πετύχουν υποστήριξη του εκλογικού σώματο και αντιμετωπίζουν διαφορετικά μειονεκτήματα για να το πετύχουν αυτό. Δηλαδή να πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε σχέσεις με τα τοπικά κόμματα, χρειάζονται χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία, Υπάρχει πρόβλημα λόγω της φροντίδας για τα παιδιά, άρα περιορίζεται ο χρόνος να πάνε να κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία, αυτό είναι εναντίον τους. Οι γυναίκες υποψήφιες και ευρωβουλευτές πολύ συχνά όταν ήθελαν υποψήφιες τους ρωτούσαν στο κόμμα πώς θα συμφιλιώσετε την πολιτική με την οικογενειακή ζωή. Ενώ τους άντρες υποψήφιους ή ευρωβουλευτές δεν τους ρωτούσαν κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια γενική τάση επανεκλογής, ε, ε, επανεπιλογής υποψηφίων παλαιών στη λίστα. Άρα είδαμε ότι έτσι μειωνόταν οι πιθανότητες οι γυναίκες να, είναι, να έχουν προτεραιότητα στη λίστα. Ευχαριστώ. Thank you. You have the floor. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για να μιλήσετε. Υποβάλλετε ερωτήσεις. Uh, Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σου. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Εγώ δεν θα σε ενταμεία της ε, παρουσιάσεις για ορισμένες επιλεγμένες χώρες και υπάρχει αυτός ο τίτλος ε, των εξαρτιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, ισορροπία μεταξύ των φύλων εάν ε, το διαβάσει κανείς ε, επιτροχάδιν, ε, διαπιστώνει το συζήτημα, είναι σοβαρό. Σχεδόν παντού οι εξαιρετίες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χαμηλή ή καμία ορατότητα. Όλα λίγο πολύ πάνε στην ίδια κατεύθυνση. Ωστόσο παρόλα αυτά τι συστήνεται δηλαδή να επικεντρωθούμε μέσω των εθνικών δραστηριοτήτων, ούτω ώστε να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών. Θα ήθελα να μας κάνετε μια περισσότερο εις βάθος ανάλυση. Βεβαίως, σαν πράγματι ότι υπάρχει χαμηλή ερατότητα αυτών των ε, πανευρωπαϊκών εκστρατιών. Ε, σε ορισμένε περιπτώσει υπήρξε κάποια ορατότητα, αλλά αυτό δεν έκανε καμία ουσιαστική διαφορά εν σχέση με τα πολιτικά κόμματα. Είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει μέσω πολιτικών ομάδων ή ε, θα έπρεπε να παρατηρηθούν τα εθνικά κόμματα να κάνουν κάποια πράγματα και να λάβουν κάποια μέτρα να βελτιώσουν την ισορροπία των φύλων. Βεβαίω η απόφαση ε, τοποθετείται σε εθνικό επίπεδο, επίπεδο κομμάτων. Γι' αυτό η σύστασή μας είναι εντός της, ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων να προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν περισσότερη επιρροή σε αυτό που κάνουν τα κόμματα σε εθνικό επίπεδο. Και η εξαρτια 50 50-50 δεν ε, χρωματοδοτήθηκε επαρκώς ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της. Και η κάλυψη εκ μέρους των ΜΜΕ ήταν πολύ μικρή. Εάν θα πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια εκστρατεία, θα πρέπει να γίνει αυτό ή δυνατόν πολύ νωρίς. Θα, θα πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις αυτές σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της προεκλογικής εκστρατείας. Ε, Νίμπλερ, ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας θα ήθελα να μας να αναφερθώ σε κάτι το οποίο εσείς κατ' δεν αναφέρετε. Ε, πραγματικά ε, έχουν ε, γραφτεί τόνοι πάνω στο θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε όλα τα επιχειρήματα. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο στο εθνικό επίπεδο. Είναι ότι όσο πιο σημαντικό θεσμικό θεωρείται το θεσμικό ε, όργανο, τόσο λιγότερες γυναίκες εκλέγονται. Και είναι ενδιαφέρον ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω το ποσοστό των γυναικών είναι 35%. Υπάρχουν κάποια εθνικά κοινοβούλια που τα ποσοστά αυτά είναι ψηλότερα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Βρετανία όπου είναι 20%, χαμηλότερο δηλαδή. Ε, ποια είναι εδώ η στατιστική συνάφεια και δεν νομίζω ότι είναι μια σύμπτωση το γεγονό ότι στη Μεγάλη Βρετανία ε, είναι αυτά τα ποσοστά. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση με τα, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι είναι ένα ε, θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Απάντηση. Ε, ναι, έχετε δίκιο. Δεν είναι τόσο επιθυμητό να εκλεγεί κανείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτιμάται το Εθνικό Κοινοβούλιο στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση τη Μάλτα, όπου είναι πολύ επιθυμητές οι σχέσεις αυτές, η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπου τα ποσοστά των γυναικών ε, είναι υψηλά και θεωρούν, ε, θεωρείται ότι είναι πολύ σημαντικό και ίσως ε, τα εμπόδια για την είσοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι λιγότερα στην περίπτωση αυτή. Ε, ε, το ποια, το πιο θεσμικό όργανο θεωρείται πραγματικά σημαντικό και πώς προσλαμβάνεται από τους υποψηφίους είναι μια καθοριστική παράμετρος. Έχετε δίκιο. Ε, ε, όπως είπε η Μέρη, αυτό είναι κάτι το οποίο μας αφορά πάρα πολύ μας τους εργατικούς, όπου το 5% είναι γυναίκες. Αλλά διαφέρει πολύ από αυτό δεν είχα την ευκαιρία να ε, διαβάσω την μελέτη σας, θα το κάνω όμως. Και διαρωτώ με κατά πόσο κάνατε αυτή την εργασία ε, όσον αφορά την εκλογή των ε, ευρωβουλευτών σε σχέση με την εκλογή πολιτικών στις χώρες που εξετάσατε. Ε, και τι γίνεται με τα ποσοστά, αν υπάρχει διαφορά στα ποσοστά μεταξύ ευρωβουλευτών και βουλευτών σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το φύλλο. Ένας από τους λόγους που είναι τόσο πολλές ε, γυναίκες ε, στην, στη Βρετανία είναι το γεγονός ότι έχουμε μια πολιτική με ένα ανώτατο όριο. Άρα λοιπόν η πρώιμη ε, παρέμβαση, η πρώιμη εκστρατεία ε, έχει σημαντικό ρόλο όπως είπατε. Πρόεδρος. Αν δούμε την περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, οι υποψήφοι θα πρέπει να είναι για να επιλεγούν και τα πράγματα είναι δύσκολα. Βεβαίω είναι πολύ δύσκολο να υποβάλει κανείς υποψηφιότητα ακόμα και σε εθνικό επίπεδο γιατί χρειάζονται πολλά χρήματα και πολλή επένδυση σε χρόνο για να κάνει κανείς την προεκλογική εκστρατεία και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να προσελκυστούν καταρχήν οι υποψήφοι, να πιστούν για να υποβάλουν υποψήφιες, να υποβάλουν υποψηφιότητα. Ε, δεν κάναμε σύγκριση ποσοστών μεταξύ ευρωβουλευτών και εθνικών ε, πολιτικών. Ε, αλλά θα συμφωνούσα με την Άννα Μπέλ ότι υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά ευρωβουλευτών γυναικών από ότι γυναικών σε εθνικό επίπεδο, γυναικών βουλευτών σε εθνικό επίπεδο. Κυρία Σούκοβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι κατανοήσαμε ότι οι ποσοστώσεις συμβάλλουν θετικά στην ε, ισότητα των ε, γυναικών ε, όσον αφορά την ε, επιτυχία των γυναικών υποψηφίων στις ε, εκλογές, ευρωεκλογές. Το κατανοώ, αλλά πιστεύω ότι ε, ότι το σύστημα αυτό, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι αρκετά βιώσιμος. Ναι, μεν έχει πρόθεσμα μια επιτυχία, Εγώ υποστηρίζω τις γυναίκες, ε, την είσοδο των γυναικών στην πολιτική, στο δικό μου πολιτικό κόμμα. Δημιούργησα το κίνημα για την συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Αλλά δεν είμαι υπέρ της εισόδου ενός συστήματος ε, ποσοστώσεων στο νόμο. Να το προβλέπει δηλαδή η νομοθεσία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, ποσοστώσεις στο εσωτερικό εντός των ε, πολιτικών κομμάτων. Δεν είχα εγώ την ευκαιρία να μελετήσω ε, τα αποτελέσματα, αλλά δεν ξέρω αν κάνετε αυτή τη διάκριση μεταξύ των ποσοστώσεων που προβλέπει ο νόμος και των εσωτερικών ποσοστώσεων που προβλέπουν τα ίδια τα πολιτικά κόμματα. Γιατί στη Σλοβακία, για παράδειγμα, υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές ποσοστώσεις των πολιτικών κομμάτων. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια φυσική αντίδραση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, τα οποία διαπιστώνουν ότι για τους ψηφοφόρους ε, είναι ενδιαφέρουσα η, συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Όλο και περισσότερο λοιπόν ε, τα πολιτικά κόμματα από μόνα τους ε, παροτρύνουν, θαρρύνουν τις γυναίκες να συμπεριληφθούν στις λίστες τους. Αυτή είναι η δική μου γνώμη τουλάχιστον. Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα το ότι είπατε ακριβώς. Θέλετε να απαντήσω στο σχόλιο σας ε, εν σχέση με την σύγκριση, την αντίστοιξη μεταξύ ε, ε, προβλέπει ο νόμος και εσωτερικών προστόσων που προβλέπουν τα κόμματα. Απάντηση. Ναι, κάναμε, το εξετάσαμε, αλλά δεν βρήκαμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα του ενός ή του άλλου αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι τα κόμματα δεν είναι αυτό, αυτά καθ' αυτά ε, υποχρεωμένα ε, να προβλέπουν ποσοστώσεις. Βεβαίως θα μπορούσαν να παροτρινθούν να συμπεριλάβουν ε, ποσοστώσεις. Μπορούν βεβαίως να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές αυτές οι ποσοστώσεις εντός των κομμάτων, εξίσου με αυτέ που προβλέπει ο νόμος. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η διάκριση. Ευχαριστώ. Εγώ θα είχα από τη δική μου πλευρά δύο ερωτήσεις που συνδέονται κάπως με το θέμα των ιστορικών ποσοστώσεων των κομμάτων ή των ποσοστώσεων που προβλέπει ο νόμος. Ποιες είναι οι σταδιοδρομίες των γυναικών που υποβάλλουν υποψηφιότητας. Είπατε ότι συχνά δεν επωφελούνται οι γυναίκες από ε, την κομματική δομή, δηλαδή τα κόμματα δεν υποστηρίζουν κατά την γυναίκε που έχουν συμπεριλάβει στη λίστα τους. Ε, βλέπετε κάποια διασύνδεση μεταξύ της προστορία μιας γυναίκας και της ε, ε, επιτυχίας, ε, της πιθανότητας να εκλεγεί. Υπάρχουν ε, επιπτώσεις στη συνολική λίστα Δηλαδή το να έχει μία γυναίκα ε, ενεργό θέση, το να έχει ένα κόμμα μάλλον, συγγνώμη, ενεργό θέση, να είναι πεπισμένο για την αξία της ε, προσπάθειας εξίσωσης των ε, φύλων προσφέρουν καλύτερες πιθανότητες τελικά στο να εκλεγούν οι γυναίκες ή όχι. Δεύτερον, βλέπετε της πιθανότητας μιας γυναίκα, η οποία ήδη εξελέγει το 2009 και υποβάλλει ψηφιότητα στο 2014, δηλαδή έχει μια σταδιοδρομία ήδη ε, στο σώμα, αυτό αυξάνει τις πιθανότητες της. Υπάρχει αυτού του είδους η συνέχεια, αν θέλετε, στις, ε, στην ε, σταδιοδρομία και στις πιθανότητες εκλογής. Απάντηση. Ε, κατά πόσο ο κομματικός μηχανισμός στηρίζει τις γυναικές υποψηφιότητες. Αυτό είναι ε, δύσκολο ακριβώς, δύσκολο να το εξετάσουμε. Ε, βλέπουμε βεβαίως ποια είναι η θέση στη λίστα και βεβαίως εάν κάποιες γυναίκες ευνοούνται έχουν περισσότερες πιθανότητες να μπουν στην κορυφή της λίστας και αυτό βεβαίως έχει μια θετική επίπτωση, ένα θετικό αντίκτυπο στις ε, πιθανότητες των γυναικών να εκλεγούν οποιοδήποτε υποψηφίου. Ε, το να είναι κανείς δηλαδή στην ε, αρχή της λίστας, στην κορφή της λίστας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ακούσαμε πολλά στις ε, συνεντεύξεις σε σχέση με το πώς ένας ευνεμένος υποψήφιος που πολύ συχνά είναι άνδρας γιατί έχει μια μακρά πολιτική προϊστορία καμιά φορά αυτοί οι υποψήφοι προωθούνται και τελικά υποτιμώνται άλλοι υποψήφοι οι όμως έχουν επενδύσει πολλά σε αυτή την εκστρατεία. Βεβαίω, ο στόχος ενός κόμματος είναι να πάρει έδρα, έδρες και θα προωθήσουν τους τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ψηφιστούν. Και αυτό είναι ένα στοιχείο του να ε, επιβραβεύουν, αν θέλετε, την ε, πίστη προς την πολιτική ομάδα. Υπάρχει, ε, πολύ συχνά είπαμε ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο δημοφιλείς από τους άντρες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μία ε, τάση αναστολής των γυναικών υποψηφίων. So you were asking about whether or not if, a woman is more experienced. Σε αυτό το θέμα της ε, προηγούμενης ε, δρέωσης μιας γυναίκας υποψηφίου στην πολιτική ζωή. Αυτό ισχύει τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. Θα ήθελα να ρωτήσω για τις κλειστές λίστες που έχουμε και που κατ' δεν ε, λειτουργούν. Όταν κάποιος ε, ψηφίζει ένα πολιτικό κόμμα, θεωρώ ότι αυτό δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Δεν θεωρώ ότι είναι μια σωστή εκλογική πρακτική να υπάρχουν ε, κλειστοί, κλειστές εκλογικές ε, λίστες. Ίσως ε, υπάρχει η πρόκληση για μας είναι να βρούμε ένα πιο δημοκρατικό τρόπο ε, ενίσχυσης προώθησης ε, των γυναικών για να διατηρήσουμε ή να βελτιώσουμε τον αριθμό των γυναικών υποψηφίων. Οι ποσοστώσεις ε, προφανώς δουλεύουν αλλά χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα για να τα εξασφαλίσουμε. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το εργατικό κόμμα αυτή τη φορά δεν ε, είχαν ε, ε, αυτή τη φορά το ποστό των γυναικών είχε ήταν το ελάχιστο δυνατό. Και πραγματικά υπάρχει μια πραγματική τάση να κάνει κανείς μόνο αυτό που πρέπει και όχι τίποτα παραπάνω. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και αν υπάρχει αυτό το σύστημα που λειτουργεί, τότε να βεβαιώσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με δική μας δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να κλείσουμε και είμαστε στη διάθεσή σας.